Με βάση τα πρακτικά και τα κείμενα που, ε, που συμφωνήσαμε, ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει επί των πρακτικών τη προηγούμενη Ολομέλεια. Οι αρχέ του ΗΠΑ